Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την ημερησία διάταξη. Στις 10 και 15 έχει προβλεφθεί να γίνει μια συζήτηση για την Τουρκία. Ελπίζω ότι θα έχουν κάποιοι συνάδελφοι αυτό μετά από αίτηση πολλών συναδέλφων. Δεν έχετε για την μέση διάταξη κάποιες ε, παρατηρήσεις. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Όχι. Έχω μία ανακοίνωση ακόμα να σας κάνω. Είμαι κάπως ενοχλημένος. Διότι ο ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου έκανε μια ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης, στον τύπο και είπε ότι είχα ε, αντιμετωπίσει μια δήλωση της κυρίας Κόπα η η οποία στη συνέχεια υποτίθεται ότι δόθηκε στον τύπο. Ακολούθησε. Υπήρξε λοιπόν μια επιστολή η οποία ακολούθησε και ζητήθηκε κάποιος εκπρόσωπος από το στρατόπεδο Ασράφ να συνεχθεί με την κυρία Χιμπόσκαβα. Το απέριψε αυτό και νομίζω ότι σας βρίσκω σύμφωνο σε σχέση με το θέμα αυτό. <clears throat> Επίσης, με την κυρία Χιμπάσκοβα σε άλλες, ε, και με άλλους ενδιαφερόμενους είχαμε συζητήσει αυτά που είπε η κυρία Κοπά σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση στο Ασράφ ότι δεν έχουν τηλέφωνο δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά, ε, βασικές υπηρεσίες, δεν έχουν τηλεόραση, δεν έχουν ίντερνετ. Και βρίσκω ενδιαφέρον να τονίσω ότι το στρατόπεδο Ασφάφ έχει μια έκταση 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και το, οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι εκεί γιατί υπήρξαν σύμμαχοι ενός αντίπαλου καθεστώτος. Και έχουν 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη διάθεσή τους. Wenn das 30 Kilometer Land in Sussex wäre, 30 λοιπόν τετραγωνικά χιλιόμετρα, όχι 30 χιλιόμετρα, δηλαδή ορθώνει ο πρόεδρος και φοβάμαι. Και το Ιράκ από την αρχή της δημιουργίας του στρατοπέδου Ασράφ είπε ότι πρέπει να κλείσει. Μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω ότι εδώ οι χώρες μας δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν να υπάρχει χώρος για τους πρόσφυγες στις χώρες μας. Να φέρουν ελάχιστους ε, πρόσφυγες οι χώρες μας. Και γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε μια τέτοια κατάσταση. Και δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση κατά συνέπεια. Νομίζω ότι μόνο με τον τρόπο αυτό, με το να δεχτούν οι χώρες μας πρόσφυγες από το, από το θα μπορέσει να λύσει το θέμα αυτό. Απλώς ήθελα λοιπόν να σας τα επισημάνω όλα αυτά και να υπενθυμίσω ότι στη συζήτηση με την Γιάννα Ιμπάσκοβα είπαμε το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί και με το Ιράκ και με την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στο Ιράκ. Αυτό είναι το σημαντικό, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Ιράκ, γιατί επανέρχεται η βία στο Ιράκ. Και δεν θέλουμε να μας εμποδίσει το στρατόπεδο Ασράφ για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που αναδύεται στο Ιράκ. Δεν βλέπω λοιπόν να έχετε κάποια αντίρρηση στα θέματα αυτά. Έχουμε τώρα επίσης μια πρόταση του κυρίου Φίλε που ζήτησε να γίνει μια σύντομη επίσημη συνεδρίαση στο πανηγυρική συνεδρίαση 1η Ιουλίου στο Στρασβούργο με την ευκαιρία της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα υπάρχουν εκπρόσωποι της Κομισιόν και φυσικά και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας. Είναι λοιπόν μια κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτή η πανηγυρική συνεδρίαση. Έχετε αντίρρηση? Εντάξει, ούτως έχει αποφασιστεί. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση, στην ετήσια έκθεση. Αυτό το οποίο έχω γράψει και είναι στη διαθεσή σας έχει συνταχθεί μόλις πρόσφατα και φυσικά δεν είναι ένα έτοιμο έγγραφο είναι ένα έγγραφο εν εξελίξη, εν επεξεργασία και φυσικά ο στόχος μου είναι να μπορέσω να συμπεριλάβω και τα σχόλιά σας στο, στη νέα μορφή του εγγράφου που θα έχετε την επόμε, τις επόμενες μέρες. Έχουμε κάνει ένα σφάλμα στο παρελθόν. Αυτή είναι και η εντύπωσή μου. Η... Μπορούμε να πούμε ότι και το Συμβούλιο έχει κάνει το ίδιο σφάλμα κατά ένα Κατά κάποιο τρόπο προσπάθησε να φτιάξει ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι όποιος θέλει να προσθέσει στοιχεία θα πρέπει να καταθέσει τροπολογίες. Αν θα κάποιος θεωρεί ότι το νότιο Τατζικιστάν δεν έχει αντιμετωπιστεί προσεκτικά σε αυτή την έκθεση. Προφανώς πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένες χώρες, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε στρατηγικά στοιχεία και στην αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωση έναντι των χωρών αυτών. Αυτό νομίζω ότι έχει νόημα. Δεν ξέρω αν το έχω επιτύχει στο έγγραφο αυτό που σα παρουσιάζω. Θα χαιρόμουν όμω ιδιαίτερα αν μου δώσετε τις ε, δικές σας παρατηρήσεις, ώστε εκεί που δεν υπάρχουν ε, επαρκή στοιχεία να μπορέσουν να συμπληρωθούν. Αλλά δεν νομίζω ότι εκτός των πεζευτών των αντιστοίχων χωρών δεν ενδιαφέρεται κανείς ε, για ένα τόσο ψηλό επίπεδο λεπτομέρειας. Και επομένως θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα κέρια θέματα, στα σημαντικά θέματα. Εκεί θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο βαθμό του δυνατού και αυτά θα πρέπει να εξάρουμε ιδιαίτερα στην έκθεση αυτή. και το θέμα θα πρέπει να είναι να έχουμε ένα ηγετικό ρόλο και να υποστηρίξουμε τις ε, προτεραιότητές μας και όχι να αντιμετωπίσουμε με ένα τρόπο σαν να είμαστε απικιακές δυνάμεις όλες αυτές τις χώρες. Λοιπόν αυτό είναι νομίζω το προκείμενο. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι μια συνολική προσέγγιση θα πρέπει να είναι αυτός ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε και θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης και πράγματι πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλες τις πολιτικές μας για να επιτύχουμε στρατηγικούς μας στόχους τέλος παράθεσης και συνεχίζω θα πρέπει να, να πείσουμε τις χώρες μέλη ότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο δεν μπορούμε να έχουμε μεμονωμένες αντιμετωπίσεις. Πρέπει επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργειακές επιλογές που έχουν τα κράτη-μέλη, οι οποίες πρέπει να εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είμαστε λοιπόν μαζί, είμαστε ισχυροί, άμα είμαστε μεμονωμένοι, δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι μια απλή εικόνα. Ίσως θα πρέπει να πούμε όλα αυτά ισχύουν με την εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου για να έχουμε και την υποστήριξη όλων των συναδέλφων ιδίω του Τζόφρι Φαν Όρντεν για το θέμα αυτό, να υπάρξει ένα βρετανικ... μια βρετανική αυτοεξαίρεση, ένα βρετανικό opt-out, ένα μόνιμο βρετανικό opt-out, ένα επιφυλακτικό, ένα μάλλον μερικό opt-out, λέει ο κύριος Χάουιτ. Όλοι συμφωνούν για το να υπάρξει μια μερική αυτοεξαίρεση. with Νομίζω ότι συγχρόνως θα πρέπει να επιζητήσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά για το πώς μπορούμε να συντεριάσουμε τα συμφέροντα που υπάρχουν αλλά και τις απαραίτητες επιλογές εξωτερικής πολιτικής. Πού βρίσκεται λοιπόν η σωστή συμβιβαστική λύση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να καθορίσουμε μια σωστή στρατηγική για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι το να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις πάρα πολλές στρατηγικές ε, εταιρικέ σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα τις κάνουμε όλες αυτές τις στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις που συνάπτουμε ναι συνέχεια, αλλά δεν έχουμε κάποια στατηγική για το μέλλον. Μπορεί αυτό να ικανοποιεί τις χώρες το να είναι στρατηγική μας εταίρεια, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει από το να έχουμε μια συνολική στρατηγική. Αυτό είναι από τα κυριότερα σημεία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε μια συνολική προσέγγιση, να καθορίσουμε ποια είναι τα συμφέροντά μας, ποιες είναι οι αξίες μας, που θα πρέπει να τις προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία πολιτικής που έχουμε από τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι το εμπόριο στην εξωτερική μας πολιτική και να συναρμόσουμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι συνεκτικό και το οποίο εξασφαλίζει ότι αντιμετωπίζουμε σωστά τα συμφέροντα των κρατών μελών μας. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη συνεκτικότητα μεταξύ των φιλοδοξιών μας, των πόρων μας και την ανάγκη να έχουμε ένα ηγετικό ρόλο. Και ίσως αυτό πρέπει να προέλθει και από τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Γιατί όσο πιο πολλές στατικές ε, εταιρικές σχέσεις είναι από το Συμβούλιο, τόσο πιο λίγα λεφτά δίνει. και υπάρχει και το τμήμα που αναφέρει τις καθευθύνουσες αρχές μας για ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Και εδώ μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό στην πολιτική γειτονία μας. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη την διαφοροποίηση που ανέφερε κάποτε ο κ. Σικώσκη, ότι στα ανατολικά έχουμε Ευρωπαίους γείτονες, ενώ στα νότια έχουμε γείτονες της Ευρώπης. Εκεί είναι λοιπόν η διαφορά και η διαφοροποίηση. Συνεπώς, θα ήθελα να συζητήσουμε από κοινού, αν έχετε κάποιες ιδέες, αν συμφωνείτε καταρχάς με την ουσία αυτών τα οποία είπα, έτσι ώστε η έκθεση αυτή να μην έχει φιλοδοξίες τις οποίες δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε. Δεν ξέρω συμφωνείτε εν Αν θέλετε όμως να κάνουμε αυτή την κανονική έκθεση μπορούμε να αλλάξουμε την πρότασή μου. Εγώ είμαι στην υπηρεσία σας το θέμα είναι να καταλήξουμε σε μια συνεκτική πολιτική θέση Mr. Duff. On. Ο κ. Εγώ είμαι αυτός που από την ομάδα των φιλελευθέρων θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα όπως επίσης και το έκανα πέρυσι προσβλέπω σε κάτι τέτοιο. Είναι μια σημαντική κοινοβουλευτική δραστηριότητα να προσπαθήσουμε με στρατηγικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε την προβληματική των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και τη θέση μας σαν κοινοβούλιο στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπατε σε σχέση με το ύφος και με τη δομή εγώ το γύρο του κόσμου νομίζω τον έκανε ο Τόμας Κούκ, δεν χρειάζεται να τον επαναλάβουμε. Και εμείς προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε ένα τέτοιο, μια τέτοια πιθανότητα στην πολιτική μου ομάδα. η απουσία συνοχής και η απουσία εμπιστοσύνης η οποία χαρακτηρίζει τις συζητήσεις στο Συμβούλιο είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Τα πράγματα φέτος ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι τον προηγούμενο χρόνο. Η ΚΕΠΑ φέτος υπέφερε. Και οι διαφωνίες για το Συριακό εξέθεσαν θα έλεγα με βίαιο τρόπο αυτή την ανικανότητα του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου λοιπόν καλούμεθα να εκφραστούμε με μεγαλύτερο θάρρος, με πιο έντονο τρόπο και να κατακρίνουμε την ανικανότητα των εκπροσώπων των κρατών μελών, την ανικανότητα των ίδιων των κρατών μελών να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με σοβαρό τρόπο αυτό που είναι η υποχρέωσή τους, δηλαδή μια κοινή πολιτική στα θέματα αυτά. Εγώ βέβαια μόλις τώρα είδα την πρόταση, το πρώτο αυτό κείμενο και γι' αυτό δεν θα τολμήσω να κάνω οποιοδήποτε σχολιασμό. Όμως να θέσω ένα ερώτημα, γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο να βγαίνει από το κείμενο που έχω μπροστά μου. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το θέμα της διεύρυνσης, για την πολιτική της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ειδικό τμήμα για την διεύρυνση. Και παρά το ότι Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια άμεση θα έλεγα προθεσμία σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη. Αυτό δεν είναι λόγος για τον οποίο δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε την μακροπρόθεσμη ανάγκη για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Um, Ευχαριστώ. Δεν θα σχολιάσω τις προηγούμενες παρατηρήσεις σας, Πρόεδρε. Ε, φυσικά αποδέχομαι ευνοϊκά αυτά τα οποία είπατε σχετικά με το θετικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέραν τούτου, χρειάζεται μια ρεαλιστική αντιμετώπιση η οποία θα δείξει ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άλλωστε είναι και η φιλόδοξη αν θέλετε προσπάθεια για την οποία όλοι εργαζόμαστε. Απαιτείται ο μέγιστος βαθμός συμφωνίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρξει μια συνεργασία. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό απαιτούμε ε, απαιτείται μάλλον να λειτουργήσει σωστά η τεράστια αυτή αρχιτεκτονική ε, της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ίσως να χρειαζόμαστε άλλωστε στον τομέα αυτό και μία κάπως πιο μετριασμένη και μικρότερη υπηρεσία εξωτερικής δράσης που να αντικατοπτρίζει την οικονομική συγκυρία. Mr. Gala. κύριος Δεν ζήτησα το λόγο, αλλά εφόσον τίθεται το θέμα, εγώ συμφωνώ με την τάση αυτή που λέτε ότι δεν πρέπει να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό οδηγό για τον πλανήτη μας, αλλά να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα σημεία έμφασης και τη διάρθρωση της πολιτικής μας, να τονίσουμε ποια είναι τα στρατηγικά μας συμφέροντα και έτσι να αντανακλάται η στάση μας στην έκθεση. Αυτό έχω να πω μονάχα. Καταρχήν θέλω να υποστηρίξω τη γενική σας κατεύθυνση. Uh, Ο κύριος Χάουιτ, νομίζω ότι αυτό που είπατε ότι δεν πρέπει να γίνει ένας κατάλογος χωρών Πρέπει να θυμόσαστε όλοι ότι αυτή ήταν η κατεύθυνση παλιά για την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο παρελθόν και εδώ και πολύ καιρό έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση και να κάνουμε αυτό το οποίο προτείνεται για την ε, τωρινή έκθεση. Αυτό ήταν ένα επιτυχές εγχείρημα, αλλά από... αποτελεί προαπαιτούμενο τα μέλη της Επιτροπής μας να δείξουν κάποια αυτοσυγκράτηση και κάποια πειθαρχία και πρέπει ο εισηγητής και οι πολιτικές ομάδες να προσπαθήσουν να αποτρέψουν το να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν ένα κατάλογο. Χρειάζεται κατάλογο χωρών. Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουν μια πειθαρχία και εγώ θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου στη δική σας προσέγγιση σε αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ πρόεδρε σχετικά με την ερώτησή σας. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την πρότασή σας. Δηλαδή, όσο και αν είναι δύσκολο, περίπλοκο και απαιτητικό, πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα στρατηγική σημασία έγγραφο. Τέτοιου είδου εκθέσεις που έρχονται από το Συμβούλιο θα μπορούσαν να συμπεριληφθεί στο βασικό έγγραφο ορίζει την στρατηγική. Αυτή όμως λείπει. Είναι σαν ένας κατάλογος με περιοχές, χώρες, γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μέσα στη χρονιά. Και δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας. Συνεπώς, εγώ στηρίζω τη δικιά σας προσέγγιση απέναντι στο θέμα και νομίζω ότι όλοι πρέπει να καθίσουμε και να προβληματιστούμε πολύ περισσότερο σε βάθος για το πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Γιατί δεν είμαι πεπισμένος ότι κάνουν πραγματικά τη δουλειά την οποία εμείς περιμένουμε να κάνουν. Και η πραγματική συνεισφορά στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχει. ας μην αφήσουμε να περάσει πάρα πολλής χρόνος, πάντως υποστηρίζω απόλυτα τη δουλειά αυτή πάνω στο έγγραφο που θα εντοπίσει στρατηγική σημασίας θέματα και υποθέσεις που έχουν μεγάλη σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κανένας άλλος δεν θέλει το λόγο από ό,τι βλέπω. Ας κάνω και εγώ τώρα κάποιες παρατηρήσεις. Λοιπόν, είναι ενθαρρυντικά αυτά που μου λέτε. Εγώ θα κοιτάξω περισσότερο να ενισχύσω αυτά που είπα στην αρχή, στο σχέδιο. Εφόσον υπάρχει συμφωνία για την προσέγγιση μου, αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Και μετά θα ήταν χρήσιμο να συζητήσουμε. Αντρίου, η διεύρυνση δεν είναι κάτι που ξεχάσαμε, αλλά εμείς ασχολούμαστε περισσότερο με την ΚΕΠΑ, έτσι. Είναι θέμα διάστασης βέβαια της εξωτερικής πολιτικής και της διεύρυνσης. Πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, τη δυναμώνει την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Υπό αυτή την έννοια θα συμφωνήσω μαζί σου και θα το συμπεριλάβω. Ο κύριος Φανόρδεν. Έφυγε. Ε, τότε θα του στείλουμε το άρθρο 24, σημείο 3 της συνθήκης, να το διαβάσει. Η πρόταση αυτή πρέπει να μπει στην ε, έκθεση ως τίτλος τι λέει. Λέει ότι τα κράτη μέλη θα στηρίξουν την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια ενεργά σε πνεύμα ε, πίστης και θα συμμορφωθούν στους, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να μην το βάλουμε αυτό στην αρχή μπροστά, στον τίτλο, τίτλος, υπότιτλος τέλος πάντων, που είναι κομμάτι από τη συνθήκη, γιατί όχι. Ο κύριος Φανόρντεν μερικές φορές έχει καλές ιδέες, πράγματι. Πιστεύω λοιπόν. Α, η κυρία Ματιματίνη. Όχι, δεν θέλετε το λόγο. Θα ενημερώσω τον κύριο Φανόρντεν για αυτό που είπατε. Δεν, ε, δεν έχω φωνή βλέπετε, οπότε δεν μπορώ να σας μιλήσω περισσότερο. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον συνάδελφο. Όλοι έχουν φωνή. Έτσι, ακόμα και αν είναι λίγο σπασμένοι. Καλώς. Τελειώσαμε με αυτό. Συνεπώς τότε. Περνάμε στον κύριο Κάσμαν. Είναι εδώ ο κύριος Κάσμαν. Πού είσαι. Εδώ. Ωραία. Παρακαλώ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Έλμερ, πρόκειται για μια ενημέρωση στην Επιτροπή μας σχετικά με την συνέργεια και τη συνεργασία που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες οι οποίες επιτελούν έργο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που είπατε για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, είχαν αρκετά μεγάλη σημασία για μένα εγώ συνάντησα τους εκπροσώπους ε, ε, αυτής της υπηρεσίας στην Νότιο Αφρική. Τους ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας εκεί και πώς αντιμετώπισαν κάποια διπλωματικά προβλήματα και επίσης και την γραμματεία τους εδώ στις Βεξέλλες. Αντιμετωπίσαμε λοιπόν ορισμένες δυσκολίες εμείς στην αρχή θέλαμε να κάνουμε μια πλήρη διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στην Νότια Αφρική, λόγω όμως των αλλαγών που επιβλήθησαν στις αντιπροσωπείες, κατά της επιθυμίας μου ως προέδρο της διάσκεψης των προέδρων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών, έχουμε περιορισμού σε σχέση με τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, ε, τις οποίες μπορούμε να στείλουμε και γι' αυτό κάναμε μια ομάδα εργασίας μαζί με τον Σαρτζεντίνη και έναν άλλο συνάδελφο Λοιπόν, πέντε μέρες πριν από την αρχή της ε, συνεδρίασης, ο συμπρόεδρος μου στη Νότια Αφρική ε, ακύρωσε ο ομόλογός μου την επίσκεψή μας. Λόγω του ότι υπήρχε υποτίθεται ε, μία παρανόηση γιατί εμείς υποβιβάζαμε την σημασία της Νοτιού Αφρικής γιατί δεν κάναμε μία πλήρη διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Αυτός είναι ο κίνδυνος ε, τον, για τον οποίο είχα προειδοποιήσει και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο συνέβη. Παρά τις συζητήσεις που είχα με την Πρόεδρο, την ομόλογό μου, ε, επέμεινε ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια δυνατότητα για άλλου τύπου συνάντηση. Ε, και χάρη στην παρέμβαση λοιπόν του Προέδρου Σούλτς, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον Μαξιζούλου, και άλλαξε επιτέλους η απόφαση αυτή και έτσι μπορέσαμε να κάνουμε την επίσκεψη και τη συνάντηση. Ήταν σαφές ότι σε τέσσερα χρόνια, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της νοτιοαφρικανικής πλευράς, μέσα σε τέσσερα χρόνια έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή θα έλεγα και σωστά εδρεωμένη μορφή συνεργασίας. Και γι' αυτό και η διάσκεψη των Προέδρων ε, με την απόφασή της ε, νομίζω ότι έβλαψε αυτήν την συνεργασία. Εν πάση περιπτώσει <clears throat> πρέπει να συζητηθεί αυτό το σημαντικό συμβάν, το θέμα της ακύρωσης που απεφεύχθη βέβαια της συνάντησης. Αυτό δείχνει τη σοβαρότητα των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την απόφαση της διάσκεψης των Πρόεδρων. Εν πάση περιπτώσει όπως είπα οι συναντήσεις έγιναν. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις και στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας και στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το εμπόριο, οι Νότιο Αφρικανοί δεν ήθελαν τα θέματα αυτά να συζητηθούν, το τελευταίο θέμα μάλλον, είχαν ανησυχίες επίσης και για τον κρατικό νόμο ε, για την ενημέρωση και τα μέσα ενημέρωσης αλλά βρήκαμε ένα κομψό τρόπο να εισάγουμε το θέμα αυτό στις συζητήσεις μας χωρίς να το έχουμε στην επίσημη μερίσια διάταξη. Φτάσαμε εκεί στο τέλος μιας πολύ σημαντικής διάσκεψης των BRIC στο Ντέρμπαν και ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενό της όπως σας είπα συζητήσαμε και το θέμα του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης που ενδιαφέρει και ανησυχεί πάρα πολύ τους εκδότες, τους καναλάρχες, ε, τα μέσα ενημέρωσης ε, και περιμένουν να δουν αν ο πρόεδρος Ζούμα θα υπογράψει το διάταγμα αυτό, το νόμο αυτό, εφόσον βέβαια περάσει από την εξέταση του συνταγματικού δικαστηρίου. Ε, τέθηκε βεβαίως και αυτό ήθελαν πολλοί να συζητηθεί η Νοτιοαφρικανή ήταν η αναπτυξιακή βοήθεια και σε σχέση με τις πιθανότητες κατάργησης της βοήθειας αυτής σε χώρες μεσαίου εισοδήματος. Έτσι φαίνεται να είναι η Νότια Αφρική αν δείτε το ΑΕΠ. Αλλά παρόλα αυτά η διαφορά ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους είναι ίσως η μεγαλύτερη στον κόσμο. Συνεπώς λοιπόν συμφωνήσαμε μαζί τους και συζητήσαμε το αν υπάρξει ένα κλείσιμο αυτής της βοήθειας της κοινοτικής στη συγκεκριμένη φάση, σε μεταβατική περίοδο για τη χώρα, θα ήταν ακατάλληλο. Κρίμα που δεν είναι εδώ ο κύριος Βανόρντεν γιατί θα μπορούσε να μεταφέρει ε, το μήνυμα αυτό και προς την κυβέρνηση συνασπισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ ε, άσκησα κριτική ε, στην Βρετανική κυβέρνηση η οποία στις 30 Απριλίου αποφάσισε ότι θα καταργήσει από το 2015 και μετά κάθε προσπάθεια αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας με την Νότιο Αφρική γιατί δίθεν δεν το έχει ανάγκη και μπορεί να χρηματοδοτήσει πλήρως τις ανάγκες της. Αυτή είναι πολύ απογοητευτική η απόφαση και η απόφαση αυτή παρουσιάστηκε μάλιστα ε, σαν κάτι στο οποίο συμφωνούσαν και οι Νότιοαφρικανοί, κάτι το οποίο περί να σας πω ότι δεν ίσχυε. Πέραν αυτών των θεμάτων, στα πλαίσια των συζητήσεων που έγιναν, συναντηθήκαμε και με ΜΚΟ επισκεφθήκαμε κάποια προγράμματα που εξελίσσονται για να δούμε με ποιο τρόπο ε, δαπανώνται τα κοινοτικά χρήματα. Με λαμπρό τρόπο χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά. Χρηματοδοτούμε ζωτικής ανάγκης προγράμματα στον τομέα της υγείας και της υγιεινής, όπως επίσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και της αηφορίας. Επισκεφθήκαμε επίσης ε, και το πρόγραμμα ίσης ε, ισότιμης ανάπτυξης ανδρών γυναικών στην πόλη της Καιλίσσα και εκεί τα κοινοτικά χρήματα παράγουν αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή προστιθέμενη αξία. Η συνεισφορά μας στον προϋπολογισμό της, της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης δεν ξεπερνά το 1% αλλά το 1 αυτό της 100 λειτουργεί σαν προστιθέμενη αξία. Και ένα πρόγραμμα το οποίο επιτυγχάνει τότε συνεχίζεται στο μέλλον με χρηματοδότηση ίδια αυτή τη φορά από τη συγκεκριμένη χώρα. Είχαμε λοιπόν μια καλή συζήτηση με ένα think tank για την νοτιοαφρικανική οικονομία. Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας προς τις υπόλοιπες χώρες της Αφρικής και ο μεγαλύτερος αφρικανός εξαγωγέας προς την Ασία όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα τα οποία σωρεύονται και είναι σοβαρά. Είχαμε επίσης και με εκπροσώπους του Εργατικού Κόμματος, ε, με τα συνδικάτα μάλλον, η συζήτηση δεν ήταν ακριβώς συζήτηση ε, πολιτική, αλλά ε, βασικά τα συνδικάτα μας είπαν ότι η απεικιοκρατία ήταν πάρα πολύ κακό πράγμα και η Κίνα είναι πάρα πολύ καλό πράγμα και δεν έχει σχέση με τις ευρωπαϊκές ε, απεικιοκρατικές χώρες. Εγώ με διπλωματικό τρόπο προσπάθησα να πω στους συνδικαλιστές ότι ε, δεν μπορούσαν να μαντέψουν ε, το τι πιστεύουμε εμείς και ότι εμείς δεν πήγαμε στην Νότια Αφρική για να μας κάνουν, ε, να μας κάνουν Και ε, στο τέλος αφού μας έκανε κήρυγμα μας χαιρέτησε λέγοντας «Γεια σας σύντροφοι» και θέλει να μας ξαναδεί. Ε, εν πάση περιπτώσει εκτός αυτού οι συζητήσεις ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν μια συνάντηση η οποία θα ακολουθηθεί από μια επίσκεψη του κυρίου Σούλτς αν δεν κάνω λάθος Προβλέπεται επίσης και μία επίσκεψη του Προέδρου στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και θέλουμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για να είναι επιτυχημένη η επίσκεψη αυτή. Αλλά αυτοί οι οποίοι δούλεψαν πολύ καλά είναι η γραμματεία της Επιτροπής και το γραφείο μου το πολιτικό που ξεπέρασαν τα εμπόδια και έγινε αυτή η συνάντηση με επιτυχία ελπίζω. Ελπίζω λοιπόν να ενθαρρύνω την διάσκεψη των Προέδρων έτσι ώστε να αλλάξει την απόφαση που πήρε σχετικά με τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες. Εγώ τους πρότεινα ο ίδιος ένα μηχανισμό μέσα του οποίου θα μπορούσαν να μειώσουν κατά το 1 τρίτο τον προϋπολογισμό και να διατηρήσουν ε, τον αριθμό των αντιπροσωπιών. Αυτοί μόνο μείωσαν τον αριθμό των αντιπροσωπιών, των αποστολών, τίποτα άλλο. Ελπίζω να αλλάξει η κατάσταση. Έλμερ δεν θα πω κάτι άλλο. Uh, uh, λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση της Επιτροπής. Ευχαριστώ, λέει ο <clears throat> πρόεδρος, χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να λάβω το λόγο στην συντομία γιατί πρέπει να πάω σε μια άλλη συνεδρία Ευχαριστούμε για την έκθεση λέει ο Σκάλερ, και για το γεγονός ότι μας δώσατε και μια πολύ καλή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην Νότια Αφρική. Είναι πολύ χρήσιμο να καταγραφεί το γεγονός ότι κάνουμε όλα αυτά στην χώρα αυτή στα πλαίσια της ανάπτυξης και της συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει η εντύπωση ότι θέλουν να μας δώσουν ορισμένα μηνύματα και να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι. Θεωρείτε ότι όλα αυτά προκύπτουν και από το γεγονός ότι σε εσωτερικό επίπεδο υπάρχει σημαντική πίεση από τα μέσα ενημέρωσης γιατί υπάρχουν πολλά σκάνδαλα και υπάρχει η συζήτηση αυτή σε σχέση με τη στάση της κυβέρνησης ότι δηλαδή χρησιμοποιούν το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουν να βάλουν κατά μέρο τα εσωτερικά τους προβλήματα που είναι λαβή για επικρίσεις και γι' αυτό έχουν κάπως επιφερειακή στάση να της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Μάικελ. Νομίζω ότι η πολιτική αντίδραση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντανακλά τη συνολική εικόνα που έχουν συλλογικά οι Νοτιοαφρικανοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πολύ σημαντικοί για αυτούς. Είμαστε ο στρατηγικός τους εταίρος. Έχουμε μια στρατηγική σχέση μαζί τους. Και είμαστε ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Νότιας Αφρικής. Περίπου 30% από το συνολικό εμπόριο της Νότιας Αφρικής ε, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από ότι με τις άλλες χώρες BRICS. Αλλά όπως μπορεί κανείς να περιμένει, μετά από τον αγώνα εναντίον του Απαρχάιτ υπάρχει ένας ιεραρχικού χαρακτήρα αγώνας. Από τη στιγμή που έχουν ληφθεί οι αποφάσεις αυτές, σιγά σιγά αυτό κατασταλάζει. Όταν περάσαμε στη δομή μιας ομάδος εργασίας, υπάρχει μια ψυχολογία που λέει όχι αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, πρέπει να το φέρουμε στα ύπατα επίπεδα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα και όπως είπατε οι εσωτερικές ε, αντιφάσεις και συγκρούσεις μέσα στο Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο επηρεάζουν τις σχέσεις μας. Και υπάρχει και μια εσωτερική διαμάχη μέσα στο κόμμα αυτό λόγω της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων που πλησιάζει το 45%. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα μέσα στην Νότια Αφρική, το θέμα των ορυχείων μαρικών, παραδείγματος χάρη. Και γι' αυτό μερικές φορές υπάρχει μια αντιμετώπιση, λες και είναι σε πολιορκία η Νότια Αφρική. Αλλά τους είπαμε και πάλι ότι έχουμε την εντύπωση ότι για σας δεν μετράει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε εκεί να αλλάζουν αμέσως αντιμετώπιση, τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής μας σχέσης. Και νομίζω ότι η επίσκεψη του Επιτρόπου το επιβεβαίωσε αυτό. Αλλά έχετε δίκιο ότι υπάρχουν εσωτερικές ε, συγκρούσεις μέσα στην Νότια Αφρική. Υπάρχουν κατηγορίες κατάχρησης και διαφθοράς εναντίον της κυβέρνησης και υπάρχουν και τα θέματα αναταραχής μεταξύ των εργαζομένων, όπως είπε και ο Άντριου Ντάφ, τα ξέρουμε εμείς από τις χώρες μας, μερικές φορές οι πολιτικοί αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά σωστά και άλλες φορές κάνουμε σαν να μην υπάρχουν τα προβλήματα αυτά και ελπίζουμε ότι θα φύγουν από μόνα τους. Αλλά η Νότια Αφρική τα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα σωστά πιστεύω. Ευχαριστώ. Κύριος... Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Έρχομαι στο σημείο 6. Εμάρ Κοστέλο. Ομάδα εργασίας για την σχέση με την Παλαιστινιακή Αρχή και επίσκεψη στη Ραμάλα στις 27 Απριλίου 2 Μαΐου. Μπορείτε να κάνετε μια παρουσίαση της ε, ε, επίσκεψης αντιπροσωπείας. Παρακαλώ χωρίς μικρόφωνο. Michael, you know that it's difficult for me. okay. Hi. Good morning, Chair. Good morning. I... Eh. Ευχαριστώ, Έλμα. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα και την πρόσκληση να σας ενημερώσω για την αντιπροσωπεία τη συνάντηση στη Ραμάλα και τη Δυτική Όχθη. Η συνάντηση έγινε από τις 27 Απριλίου μέχρι τη Δευτέρα Μαΐου. Αποτελεί το η αντιπροσωπεία μας από εμέ την Ιδία, από τη Βερονίκ Ντοκεζέρ και τον Αλεξάνδρε Τάιν από τους Φιλελευθέρους, από ένα εκπρόσωπο των Πρασίνων και από τον κύριο Τούσια από την ΚΟΕ. η διάσκεψη των Προέδρων μας έδισε την δυνατότητα να πάρουμε μέρος σε μια διάσκεψη η οποία είχε οργανωθεί στη Ραμάλα πριν από την αρχή της επίσημης αντιπροσωπείας, της επίσημης επίσκεψης. Ελευθερία και αξιοπρέπεια λεγόταν η συνάντηση αυτή για τους Παλαιστινίους οι οποίοι κρατούνται στο Ισραήλ 11 χρόνια μετά από την ομιλία του ε, Μπαργκουτή και στη διάσκεψη αυτή υπήρξαν ανώτεροι διπλωμάτες από όλο τον κόσμο και αρκετοί βουλευτές και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρξαν και προηγούμενοι πρόεδροι του Παλαιστινιακού Συμβουλίου όπως ε, επίσης και πρόεδρε της αντιπροσωπείας με το Παλαιστινιακό Συμβουλίο και αναφέρομαι στην κυρία Μοργαντίνη. Είπαμε 11 χρόνια από τη σύλληψη του ε, Μαρουάν Μπαργκούτη. Το θέμα ήταν οι, οι φυλακισμένοι ε, αυτή τη στιγμή πάνω από 4.000 άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μέλη της Παλαιστινιακής Βουλής τα θέματα τα οποία τέθηκαν στη συνάντηση αυτή ήταν ε, η έλλειψη ε, κατηγοριών, οι συνθήκες κράτησης, ο θάνατος ενός μεγάλου αριθμού, η υποκράτηση Παλαιστινίων, η κράτηση γυναικών, η κράτηση παιδιών και η φυλάκιση επίσης Παλαιστινίων στο Ισραήλ, κάτι το οποίο παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τις οικογενειακές επαφές και επισκέψεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Μαρτίου ε, υιοθέτησε ένα ψήφισμα ζητώντας να υπάρξει μια επιτροπή έρευνας η οποία να εξετάσει τις συνθήκες κράτησης των Παλαιστινίων στο Ισραήλ αλλά η συμμετοχή μας στη διάσκεψη αυτή και τα θέματα τα οποία τέθηκαν απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι η ε, ε, αποστολή μιας τέτοιας συγκεκριμένης ομάδας έρευνας από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατεπηγόντως. Σχετικά με τη διάσκεψη αυτή, ελευθερία, αξιοπρέπεια, ότι υπήρξε μία συνάντηση επίσης ε, μεταξύ των Προέδρων και των εκπροσώπων του Παλαιστινιακού Συμβουλίου όπως επίσης και όλων των Προέδρων και Αντιπροέδρων των, των ε, διακοινοβουλευτικών επιτροπών με το Συμβούλιο αυτό για την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού ε, μεταξύ τους. Το πρόγραμμά μας από εκεί και πέρα ήταν ιδιαίτερα εντατικό Καταρχάς ε, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους του νομοθετικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου, συναντηθήκαμε με τον Φαγιάντ, τον προηγούμενο ε, προ, ε, πρωθυπουργό, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ολοένα πιο δύσκολη πολιτική κατάσταση μετά από την αποστολή του Κέρι στην περιοχή που θα έπρεπε να γίνει μέχρι τις 7 Ιουνίου, αν και ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο θα καθυστερήσει περισσότερο. Επισκεφθήκαμε επίσης κάποιες από τις πόλεις, κάποια από τα χωριά που βρίσκονται στην γραμμή διαχωρισμού, στην κοιλάδα του Ιορδάνη είδαμε τις συνεχείς εκενώσεις πληθυσμού οι οποίες γίνονται στην περιοχή αυτή. Ε, είδαμε επίσης ότι και λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων του Ισραηλινού στρατού έπρεπε να μετακινούνται συνεχώς, έπρεπε να κλείνουν τα σχολεία και αυτά φυσικά τα οποία συμβαίνουν είναι εντελώς απαράδεκτα πράγματα και δημιουργούν προβλήματα στη ζωή των Παλαιστινιακών κοινοτήτων. Συναντηθήκαμε επίσης και με τον, εκπρόσω, τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, μας ενημέρωσε για την πολιτική κατάσταση. Πήγαμε στο βορρά, στη Τζενίν. συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας και με εκπροσώπους του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, πήγαμε στην Ευρώνα, ε, είδαμε την ε, παλιά πόλη της Ευρώνας, είδαμε τις επιπτώσεις ε, της ασφικτικής μορφής ελέγχου του Ισραηλινού στρατού στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συναντηθήκαμε με εκπροσώπους ΜΚΟ που μας παρουσίασαν την άποψή τους για την κατάσταση την οποία βιώνουν. Τώρα για τα συμπεράσματά μας που βγήκαν από τις επισκέψεις μας και τις συναντήσεις τις οποίες είχαμε. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη έχετε διαβάσει το ανακοινωθέν τύπου το οποίο κυκλοφορήσαμε. Εκφράσαμε την ανησυχία μας, την βαθιά ανησυχία μας για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην περιοχή ε, για το πώς ε, έχουν, τους έχουν απαρνηθεί στους Παλαιστινίους εννοώ θεμελιώδη δικαιώματα, ε, την ελευθερία κίνησης καταρχάς. Όλα αυτά τα σημεία ελέγχου, τα checkpoints τους δημιουργούν τεράστια προβλήματα, χωρίζουν τις οικογένειες, απομονώνουν τις κοινότητες και είναι κάτι το εξαιρετικά οδυνηρό. Ιδιαίτερα ανατολικά της πόλης της Ιερουσαλήμ. Είδαμε επίσης και το επίπεδο γενικά ε, παρενόχλησης των Παλαιστινίων σε καθημερινή βάση Είδαμε στη συνάντηση που είχαμε με τους Βεδουίνους της κοιλάδας του Ιορδάνη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Συναντηθήκαμε με Παλαιστινίους στην Ευρώνα και σε διάφορες άλλες περιοχές και πόλεις. Βλέπουμε ότι οι έπικοι από τη μία ατιμωρητοί διώκουν και ασκούν βία εις βάρος των Παλαιστινίων ε, κατοίκων και κάποιες από τις εμπειρίες τις οποίες νιώσαμε στην ε, Ευρών όπου και εμείς οι ίδιοι υποστήκαμε παρενόχληση και από τους επίκους και από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισραηλίνας. Δυστυχώς ε, το χωροτακτικό κομμάτι ε, εξαρτάται πλήρως από τις ε, νομοθετικές ρυθμίσεις του Ισραήλ που επιτρέπουν τη συνεχή διεύρυνση των κατοικιών των επίκων, των περιοχών στις οποίες εγκαθίστανται οι έπικοι και την συστηματική συρρήκνωση των περιοχών στις οποίες κατοικούν οι παλαιοί κάτοικοι. Οι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν σε ορισμένους δρόμους, σε ορισμένες λεωφόρους, ιδιαίτερα στην Ευρώνα, όπου όπως είπα δεν περνούν από ορισμένους δρόμους, αλλά αν περνούν από τους δρόμους αυτούς θα πρέπει να κυκλοφορούν στη μία πλευρά του δρόμου. Συναντηθήκαμε επίσης και με τις ε, χριστιανικές κοινότητες προσπαθούν να αναπτύξουν επίσης και με τις, τις, τους οικονομικά υπεύθυνους της περιοχής, κάνουν κάθε προσπάθεια για να αναπτύξουν οικονομικά την περιοχή τους, αλλά δυστυχώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα, οι πρόσοδοι από τη φορολογία δεν αποδίδονται και γενικά συνεχίζουν να έχουν πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα. Έχουν προβλήματα σε σχέση με τους φυσικούς πόρους, όπως με τους υδάτινους πόρους, και υπάρχουν τεράστια προβλήματα γιατί πάρα πολλοί Παλαιστίνοι πρέπει να ταξιδεύουν ε, μεγάλες αποστάσεις για να μπορέσουν να προμηθευτούν νερό. Άποψη της αντιπροσωπείας ε, δείχνουν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο έτσι ώστε να φύγουν οι Παλαιστίνοι από τις γέες τους και να μειωθεί η Παλαιστινιακή παρουσία στην περιοχή. Αυτό κάνει και ο τείχος του διαχωρισμού στην περιοχή και αυτό είναι ένα απαράδεκτο πρόβλημα διότι οδηγεί στην παρακράτηση γεών εις βάρος των Παλαιστινίων όπως ακριβώς είχε γίνει και στις δεκαετίες του 70 και του 90 και όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά εντυπωσιαστήκαμε εν πάση περιπτώσει από τους Παλαιστινίους τους οποίους συναντήσαμε οι οποίοι ε, επιζητούν μια ειρηνική διευθέτηση, μια ειρηνική διευθέτηση στα πλαίσια της οποίας να τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτοδιάθεσης όπως και το δικαίωμα να παραμείνουν στην πατρίδα τους. Είχαν προσδοκίες υψηλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα πίεζε για να λυθεί το πρόβλημα της περιοχής θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα κινηθούμε. Συμπερασματικά και σε σχέση με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα θα υπάρξει μια επίσημη έκθεση η οποία θα είναι διαθέσιμη περίπου σε δύο εβδομάδες. Οι δηλώσεις τις οποίες εκδώσαμε κατά τη διάρκεια της συνάντησης έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Θα υπάρξει κατάθεση των εγγράφων αυτών και στην ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και στους εκπροσώπους των κρατών μελών. Θα στείλουμε επίσης την τελική έκθεση και στους εκπροσώπους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ήδη η διακοινοβουλευτική αυτή συνάντηση είπε ότι η επίλυση ε, του Παλαιστινιακού είναι πολιτική προτεραιότητα. Είχαμε επίσης μια συνάντηση και με την Λέιλα Σαχίντ και με τον Ιρλανδό Υπουργό Τζο Κοστέλο ε, και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάποια θετικά βήματα. Um, we attended the Freedom and Dignity Conference. Επίσης αναφερθήκαμε και στη συνάντηση στη Ραμάλα τον μήνα Απρίλιο. Μετά από τη συνάντηση αυτή ελευθερία και αξιοπρέπεια Υπήρξε εκπρόσωπος του Μάρτουν Σούλτς στη συνάντηση αυτή. Ο αντιπρόεδρος που είχε πάει ζήτησε, έστειλε μάλλον μία επιστολή στον Μάρτιν Σούλτς αναφερόμενος στα τεκτενόμενα κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής. Και περιμένουμε και την ανταπόκριση του Προέδρου και του Προέδρου της, ε, της Επιτροπής των Αντιπροσωπιών. Δεν έχω να πω περισσότερα γύρω από το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Κυρία Ουρκίσα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Κοστέλο, και βλέποντας και τις εκθέσεις για το γεγονός ότι είναι περίπου 5.000 οι κρατούμενοι Παλαιστίνοι στο Ισραηλινό έδαφος και τις παραβιάσεις όλων των διεθνών συμβάσεων, τις ε, συνθήκες λοιπόν κράτησης που δεν τηρούν τα ελάχιστα σε επίπεδο δικονομικών εγγύσεων, Υπάρχουν γυναίκες, παιδιά που είναι κρατούμενοι, όλα αυτά που λέει η έκθεση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Θα κάνουμε τίποτα. Θα κάνει κάτι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό που αφορά τη συνεργασία με το Ισραήλ, θα κάνουμε κάτι σε σχέση με τις συμφωνίες εμπορικών ανταλλαγών για το πρόγραμμα πλαίσιο της έρευνας. Όταν βλέπουμε ότι επικρατεί αυτή η κατάσταση, σε μια οποιαδήποτε χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέσει συνεργασία, νομίζω ότι κανονικά θα είχαμε λάβει ήδη κάποιες, ε, κάποια μέτρα, είχαμε κάνει κάποιε ενέργειε Ευχαριστώ, λέει ο Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Κοστέλο. Σα ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Οι συνθήκες κράτησης των ε, φυλακισμένων, των κρατούμενων, είναι αποτρόπαιες και νομίζω ότι είναι σαφές αυτό και από το ψήφισμά μας της 14 η Μαΐου όταν μιλήσαμε για το θάνατο Αριφά και το γεγονός ότι είναι 4.000 και πλέον κρατούμενοι κάτω από πραγματικά αποτρόπες συνθήκες. Πολλοί από αυτούς ζουν σε ανθίγινες συνθήκες, δεν έχουν καμία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και η κατάσταση είναι πραγματικά αθόρυτη. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι αποφασίσαμε ότι θέλουμε να θεσπίσουμε μια προτεραιότητα πολιτικού επίπεδου για την αντιπροσωπεία μας, τονίζοντας ιδιαίτερα το θέμα των κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές. Αν δείτε την έκθεση τώρα σε σύνολο και δείτε τις συνθήκες και τη μεταχείριση που υφίστανται οι Παλαιστίνοι και τις σημαντικές παραβιάσεις που λαμβάνουν χώρα για το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό και παραδεκτό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατάει απόσταση και να μην αναλαμβάνει καμιά δράση για τα θέματα αυτά. Εγώ θα υπεστήριζα λοιπόν απόλυτα οποιαδήποτε κίνηση η οποία θα εξασφάλιζε το ότι το Ισραήλ θεωρείται υπόλογο για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο όμως πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι απαραίτητο επίσης να δώσουμε συνέχεια και στην ερευνητική αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αναφέρεται και στο ψήφισμα της 14ης Μαρτίου γιατί ιδιαίτερα η κατάσταση των κρατουμένων Παλαιστινίων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ένας από τους πέντε, ένας σε κάθε πέντε Παλαιστινίους έχει βρεθεί κάποια στιγμή στη φυλακή. Αυτό το θέμα λοιπόν δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από άλλα προβλήματα σε άλλες πολιτικές καταστάσεις, σε άλλες χώρες του κόσμου, όπου βλέπουμε την κατάσταση των κρατουμένων. Είναι πραγματικά λυπηρό το να ξέρετε ότι κάθε οικογένεια μέσα στην, ε, στα Παλαιστινιακά εδάφη έχει κατά κάποια εποχή, σε κάποιο χρονικό διάστημα, ε, είχε σε κάποιο σημείο κάποιο μέλος οικογένειας στις φυλακές. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να προωθήσουμε μια μόνιμη λύση στα προβλήματα αυτά της Μέσης Ανατολής και υποστηρίζουμε πιο στεναρή δράση. Πρέπει να υπάρξει πιο στεναρή δράση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Δίνει το λόγο στον επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Κόβατσεφ είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εταίροι μας να σέβονται το διεθνές δίκαιο, το κράτο δικαίου και να σέβονται την αξιοπρέπεια όλων των πολιτών στην επικράτειά τους ανεξάρτητα από την εθνοτική τους προέλευση. Στην τόσο δύσκολη αυτή και ευαίσθητη κατάσταση θα πρέπει να ακούσουμε την άποψη όλων των πλευρών και αναρωτιέμαι αν συναντήσατε και Ισραηλινά θύματα τρομοκρατίας γιατί κάποιοι από τους ε, κρατουμένους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ δυστυχώς ξαναγύρισαν σε παράνομες δραστηριότητες. Και αν δούμε μοναχα τη μία πλευρά του προβλήματος, σίγουρα δεν θα βοηθήσουμε τη διαδικασία συμφιλίωσης και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ξέρω ότι υπάρχουν ευαισθησίες από όλες τις πλευρές, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην έχουμε μια καταδίκη μόνο της μίας πλευράς στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ λέω πρόεδρος. Θέλω εδώ να σας πω ότι η αντιπροσωπεία που πήγε, πήγε στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το θέμα μας ήταν οι κρατούμενοι. Συναντηθήκαμε λοιπόν με εκπροσώπους των Παλαιστινίων. Το Νοέμβριο όμως, ίσως να θυμόσαστε, ότι είχαμε μια ερευνητική αποστολή επιτόπου και επί τη ευκαιρία αυτή είχαμε επαφές με μέλη της Κνεσέτ. Και τότε συζητήσαμε διάφορα θέματα και απογοητευτήκαμε πάρα πολύ επειδή την τελευταία στιγμή ακυρώθηκε εκείνη η αποστολή. Έχετε δίκιο που λέτε ότι όταν υπάρχει μια διαμάχη, μια σύγκρουση πρέπει να διασφαλίζουμε ότι ακούμε όλες τις πλευρές. Όμως όταν ένα κράτος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλες χώρες να λένε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό. Ότι το κράτος αυτό δεν πρέπει να κάνει τέτοιες παραβιάσεις. Αντιλαμβάνομαι αυτά που λέτε. Εγώ είμαι Ιρλανδή, βλέπετε, έρχομαι κι εγώ από μια πόλη που έχει περάσει πολλά που είναι και αυτοί χωρισμένοι, αντιλαμβάνομαι και υπάρχουν μερικά κοινά. Και στην περίπτωση της Ιρλανδίας υπάρχουν διαφορετικές πλευρές και καλό είναι να ακούει κανείς όλες και τις δύο. Όταν όμως υπάρχει αδικία που γίνεται και παραβιάσεις που γίνονται από μια χώρα, αυτή η χώρα πρέπει να κατονομάζεται. Και η διεθνής κοινότητα πρέπει να πει ότι είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τρομοκρατικές ενέργειες από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, και ότι δεν πρέπει αυτές να τις καταδικάζουμε. Κάθε τρομοκρατική ενέργεια πρέπει να καταδικάζεται. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά οι Παλαιστίνοι με τους οποίους συναντηθήκαμε, όταν ακούσαμε τη δικιά τους θέση, θα έλεγα ότι πρόκειται για ειρηνικούς πολίτες, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν για μια ειρηνική λύση. Το είδαμε αυτό και είδαμε πόσο επίμονα θέλουν την ειρήνη. Νομίζω λοιπόν πάνω σε αυτήν την καλή θέληση των Παλαιστινίων πρέπει να χτίσουμε, παρόλο που έχουν να αντιμετωπίσουν φοβερές δυσκολίες. Πρόεδρος. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο. Για την Τουρκία τώρα. Είχαμε πει ότι θα συζητήσουμε. Περιμένουμε την κυρία Αλεξάνδρα Κλασκάνιεν από τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ζήτησαν να γίνει μια συζήτηση σήμερα για τις εξελίξεις στην Τουρκία. Βλέπουμε ότι από ένα Καταρχήν οικολογικό πρόβλημα, πρόβλημα χωροταξίας στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε μια γενικότερη σύγκρουση και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί έχουμε μια χώρα που είναι εταίρος, μέλος του ΝΑΤΟ, υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία έχουμε στενούς δεσμούς και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συνολική ενωτική στάση σε ό,τι αφορά την επαφή των κυβερνητικών αρχών με την κοινωνία και βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα στο επίπεδο αυτό αν δούμε το γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι συνασπίστηκαν στην ε, διαμαρτυρία αυτή. Είναι πολλοί οποίοι θέλουν να επανέλθουν στην ε, κοσμική Τουρκία του Ατατούρκ. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εμπνέονται από το παράδειγμα της Αραβικής Άνοιξης και θέλουν να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα πολιτικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κινήματα αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το ίντερνετ και ιδίως το Twitter. Και είδαμε επίσης ότι χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερη βία κατά των διαμαλτω, ε, διαμαρτυρώμενων, διαδηλωτών. Πολλοί θεωρούν ότι η αντίδραση του Πρόεδρου Αβδούλαχ Γκιούλ που είπε ότι η δημοκρατία δεν είναι μονάχα εκλογές κάθε, κάθε τέσσερα χρόνια κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να υπάρξουν ε, διαδικασίες μέσα στην τουρκική κοινωνία που να επιτρέπουν οι αντίμαχες απόψεις να ακούγονται. Εμείς βέβαια δεν κατανοούμε πλήρως την πολυπλοκότητα της κατάστασης στην Τουρκία και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο να ακούσουμε απόψεις και να πληροφορηθούμε καλύτερα για το υπόβαθρο αυτής της διαμαρτυρίας που λαμβάνει η χώρα. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι ο αναπληρωτής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Μπουλέντ Αρίνς ζήτησε συγγνώμη για την υπερβολική βία της αστυνομίας στις πρώτες μέρες, αλλά όχι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κύριος Ερδοάν. Και βλέπετε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για περαιτέρω εξέλιξη στα θέματα αυτά και αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο παραμένει. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι υποστηρίξαμε στο παρελθόν την προσπάθεια του Ερντοάν να ξεπεράσει την αντίδραση των ε, στρατηγών του στρατού και θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να μπορέσει να υπάρξει μια διαδικασία δημοκρατικοποίησης στα πλαίσια της διαδικασίας προσέγγισης της ε, Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από τη στιγμή που έχει καταφέρει να παραμερίσει την αντίδραση και την αντιπολίτευση στην Τουρκία, βλέπουμε να προωθεί τις δικές του απόψεις μια Ισλαμική προσέγγιση το ερώτημα, παραδείγματο χάρη, του, της απαγόρευσης της κατανάλωσης νεοπνευματοδών μπορεί για κάποιους συναδέλφους να μην παίζει ρόλο. Για τον κύριο Νταφ, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι ένα λεπτομεριακό θέμα στην νομοθεσία. Το γεγονός όμως ότι στην νομοθεσία παρισφρίουν οι Ισλαμιστικές τάσεις και ξεπερνούν τις προηγούμενες κοσμικές αντιμετωπίσεις, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παραγνωρίσουμε και λέει ο Ερντογάν ότι θέλει να φτιάξει τζαμί τώρα στην πλατεία Ταξίμ. Κάπου πρέπει να θέσουμε σε αντιπαράθεση όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ για την δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό Χαίρομαι για την παρουσία όλων αυτών οι οποίοι είναι παρόντες και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Κύριε Καστάνγκερ είναι παρούσα. Και μετά θα ήθελα η Ρία Όμεν, η εισηγήτριά μας για την Τουρκία, να λάβει το λόγο. Η Κομισιόν. Κύριο Σπόρτμαν για την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Είμαι σύμβουλος ε, της ε, υπάτης εκπροσώπου για τα θέματα της Τουρκίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Τουρκία είναι οι μεγαλύτερες ε, αναστατώσεις κοινωνικές τα τελευταία 11-12 χρόνια. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να το δούμε μέσα από μια κάποια προοπτική και να αποφύγουμε παραλληλισμούς εύκολους με αυτά τα οποία συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία παραμένει μια εν λειτουργία δημοκρατία. Το κόμμα ΑΚΠ έχει κερδίσει τρεις εκλογές και υποστηρίζεται από το 51% του πληθυσμού και ο κ. Σερτοάν είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός της χώρας. Το πρώτο θέμα ήταν μια περιβαλλοντική θα έλεγα διαδήλωση για την πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη. Το δεύτερο θέμα ήταν κάποιες ευρύτερες ε, διαδηλώσεις που έγιναν σε πολλές πόλεις οι οποίες έχουν λιγότερο συγκεντρωμένο θα έλεγα μήνυμα και εκφράζουν μια κάποια δυσθυμία ε, την οποία έχουν αναπτύξει λόγω της έλλειψης δυνατότητας έκφρασης στην ε, κοινοβουλευτική ε, αυτή χώρα. Και τρίτον βλέπουμε μια κυκλική έκφραση κατανάλωσης, απόρριψης μάλλον και θυμού απέναντι στις βίες πρακτικές των τουρκικών αρχών καταστολής. Τα θέματα είναι σαφή βέβαια το πρώτο από τα θέματα που έθεσα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαβούλευση και συζήτηση. Στη δεύτερη παρατήρηση είναι να υπάρξει επιμονή στην ελευθερία έκφρασης, στο σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας συγκέντρωσης και στα κοινωνικά μέσα, τα ηλεκτρονικά. Και στο τρίτο θέμα είναι η καταδίκη της υπερβολικής βίας εφόσον αποδειχθεί και μια γρήγορη και αντικειμενική εξέταση αυτού του τύπου των ισχυρισμών. Οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθε από τον Τούρκο Αντιπρόεδρο και οι συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους των συνδικάτων και με εκπροσώπους των διαδηλωτών είναι ένα θετικό βήμα. Νομίζω όμως ότι στο τέλος της ημέρας ο πρόεδρος Ερντογάν θα επιστρέψει από την επίσκεψή του στις Ηνωμένε Πολιτείε και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε το τι θα μας πει σήμερα ή αύριο. Σχετικά με τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση εξεφράστη συνεκτικά Ακούσαμε δηλώσεις και από τον Επίτροπο Φούλε και από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και οι δύο θα έλεγα πρόλαβαν τα γεγονότα ε, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εξέφρασε την ανησυχία της για την δυσανάλογη χρήση βίας. Η κυρία Ασφόρντ εξέφρασε ε, ε, τα αισθήματά της απέναντι σε αυτούς οι οποίοι τραυματίστηκαν από την αστυνομική παρέμβαση. Οι δηλώσεις της ε, κυρίας Άσφορντ παραμένουν. Παρακολουθεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης από πολύ κοντά τα θέματα αυτά σε καθημερινή βάση, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αντιπροσωπεία μας στην Άγκυρα, με τις αντιπροσωπείες των άλλων κρατών μελών που υποστήριξαν και αυτές ε, τη δήλωση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αύριο θα υπάρξει επίσης ε, μια επίσκεψη στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης από το Τουρκικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων που θα καταθέσουν μια αναφορά διαμαρτυρίας ε, σε σχέση με το τι κάνει η κυβέρνηση Εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε και τις δηλώσεις όπως είπα του Τούρκου Πρωθυπουργού ε, αύριο μάλλον. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόκ. Έχω να κάνω δήλωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, τα γεγονότα έχουν ως εξής η χρησιμοποίησε υπερβολική βία η αρχές εμβολής ε, του νόμου δηλαδή στην ε, Τουρκία απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές στην πλατεία Ταξίμ. Η διαμαρτυρία αυτή τώρα έχει διαδοθεί και έχει φτάσει και σε άλλες πόλεις. Μετά από αυτήν την απρόσμενη και μεγάλη κινητοποίηση που κατέληξε και σε απώλεια ζών, η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν προσπαθεί να έχει διάλογο και να καταλήξει σε συνένεση. Αδυναμίες δηλαδή. Επιπλέον, ομόφωνα, ο τύπος αποσιώπησε ουσιαστικά τα γεγονότα. Κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν υπάρχει ελευθερία ή υπάρχει λογοκρισία από τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης. Οι αρχές λοιπόν πρέπει να φροντίσουν να διασφαλίσουν την ελευθερία του λόγου και, του, ε, και της συγκέντρωσης των πολιτών, να φροντίσει για διάλογο και να αποκαταστήσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Η τρέχουσα κατάσταση, κατά τη γνώμη μας, επίσης αποτελεί μια ευκαιρία για την Τουρκία, προκειμένου να αντιληφθεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και την ανάγκη να φροντίσει για καλύτερες διαγραφές δημοκρατίας. Επίσης πρέπει να δώσει σημασία σε όλες τις ομάδες της κοινωνίας, ακόμα και σε εκείνους οι οποίοι νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τώρα όπως γνωρίζετε, θα γνωρίζετε μάλλον, ο Επίτροπος Φιούλε πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παρευρεθεί εκεί σε διάσκεψη για ένα νέο μέλλον της Τουρκίας και τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι είχε προβλεφθεί η συμμετοχή αυτή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ο στόχος ήταν να δώσει την άποψή του ο Επίτροπος και η Επιτροπή γενικότερα για το πώς η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να δουν ένα κοινό μέλλον μεταξύ τους. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης στην Τουρκία, ο Επίτροπος θα αναφερθεί και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τουρκία στη δημοκρατική της ζωή και γενικότερα για να ανταποκριθεί στα πολιτικά κριτήρια. Εννοείται ότι εμείς στην αντιπροσωπεία η Επιτροπή και ο Αρμόδιος Επίτροπος παρακολουθούμε από κοντά τα γεγονότα. Σας ευχαριστώ. Κυριόμεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω με το εξή. Πιστεύω πως η αντίδραση της ε, υπηρεσίας μας εξωτερικής δράσης καθυστέρησε. Την είχαμε την Κυριακή μόνο. Εγώ αλλά και ο Επίτροπος αντιδράσαμε αμέσως την Παρασκευή. Συνεπώς εκφράζω εγώ στην ε, δήλωσή μου αυτή την ανησυχία μου για την υπερβολική βία που χρησιμοποίησε η αστυνομία. Και πραγματικά οι εικόνες που είδαμε βίας ήταν σοκαριστικές. Και όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες τουρκικές πόλεις. Και δεν ε, τάραξαν μόνο εμένα, αλλά νομίζω και οποιοδήποτε άλλον εκτός Τουρκίας, αλλά και μέσα στην Τουρκία. Στα ψηφίσματά μας, Πρόεδρε, εμείς έχουμε πάντα υπογραμμίσει πόσο μεγάλη σημασία έχει για την Τουρκία να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να διασφαλίσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ιδιαίτερα την ελευθερία έκφρασης. Όπως επίσης το δικαίωμα του συναθρίζεστε, αλλά και το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι μόνο οι νομικές μεταρρυθμίσεις. Το θέμα είναι και η νοοτροπία. Και όπως και εσείς, έτσι και εγώ, είμαι πάρα πολύ απογοτευμένη από τις αντιδράσεις του Πρωθυπουργού Ερτογάν. Γιατί δεν δείχνει να νοιάζεται για τις επιπτώσεις που έχει η γλώσσα που χρησιμοποιεί η δράση της κυβέρνησης επί ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας των Τούρκων που δεν τον ψήφισαν. Πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι η δημοκρατία είναι κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να λάβει υπόψη και την θέση της μειοψηφίας. Και αυτό όχι μόνο νομικά, αλλά και ως νοοτροπία στην κοινωνία. η λέξη συμβιβασμός δεν φαίνεται να υπάρχει στην τουρκική πολιτική. Θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν η στάση και της τουρκικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαίο. Ίσως θα έπρεπε να ακούσει, όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, να ακούσει προσεκτικά αυτά που είπε ο Πρόεδρος Γκιούλ, ο οποίος είπε ότι η δημοκρατία είναι κάτι παραπάνω από εκλογές. Δεν φτάνει δηλαδή. Χρειάζεται ένα πλουραλιστικό δημοκρατικό σύστημα το οποίο να είναι ικανό και να διαθέτει και μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Το έχουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και αυτή είναι μια πρόκληση. Πρόεδρε, πολλά ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για την στάση των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία ότι δεν ανέφεραν τις ταραχές. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Ότι τα μέσα ενημέρωσης αντί να αναφέρονται για τα γεγονότα στο ταξίδι Αντί λοιπόν να δείχνουν τις εικόνες, τους καπνούς που βγαίνουν από τη λατεία ταξίμα, είχαν ένα ντοκιματέρ για Τα μέσα ενημέρωσης λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι συγκεντρωμένα και ανήκουν σε συγκεκριμένα μέσα και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Τα πρόσφατα γεγονότα λοιπόν, τα τόσο καταστροφικά, ίσως αποδειχτούν μια κρίσιμη καμπή στην όλη διαδικασία. Και αν κοιτάξετε την νομοθεσία τη σχετική με την κατανάλωση νοπνεύματος για παράδειγμα, εδώ κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Αν όμως ο κόσμος πιστεύει ότι δεν πρόκειται μόνο για την προφύλαξη αυτή, αλλά κάποιος προσπαθεί να τους αλλάξει τον τρόπο ζωής τους, αυτό θα είναι επικίνδυνο. Ελπίζω λοιπόν και οι τουρκικές αρχές να το αντιληφθούν αυτό και να πάρουν κάποιο μάθημα από την όλη αυτή ιστορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλούς οι οποίοι ζητούν το λόγο. Μπορείτε να περιοριστείτε σε 1,5 λεπτό ο καθένας, παρακαλώ. Όχι. Τότε θα σας δώσω το λόγο στο τέλος και να δούμε πόσο χρόνο θα έχουμε τότε που θα έχει απομείνει. Πρέπει να δείξουμε αυτοσυγκράτηση με συναδελφικό τρόπο. Ο κύριος Χάου είναι ο πρώτος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεχτήκατε να γίνει αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν τώρα διαμαρτυρίες σε 60 πόλεις στην Τουρκία και εδώ στην πλατεία Λουξεμβούργου υπήρξαν διαμαρτυρίες και είναι φανερό ότι ακούγεται η φωνή του μέχρι και εδώ. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο να εκφράσουν την τη μεγάλη ανησυχία τη Ευρώπη για την δυσανάλογη αντίδραση της αστυνομία και να τονίσει την ανάγκη του διαλόγου. Θα πρέπει όπω και οι ΗΠΑ να τονίσουμε ότι είναι δίκαια έκφραση δημοκρατικών δικαιωμάτων η διαμαρτυρία και θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει λογοδοσία για όλους αυτούς οι οποίοι χρησιμοποίησαν υπερβολική βία. Πρέπει επίσης να εκφράσουμε και τα συλληπιτήριά μας για τους τρεις διαδηλωτές οι οποίοι σκοτώθηκαν στις διαπραγματεύσεις. Ένας από τους οποίους είναι από την νεολαία του JHP. Οι εκατοντάδες λοιπόν των τραυματισμένων και ιδίω όλοι αυτοί που χωρίς να συμμετέχουν τραυματίστηκαν και αυτό συμβολίζεται από τη γυναίκα με τα κόκκινα που έχουμε δει στις φωτογραφίες Επίσης γνωρίζετε ότι υπήρξε μια, ε, ρίξανε δακρυγόνα στο Παξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλοί οι οποίοι εκδιώχτηκαν από τα δακρυγόνα, οι διαδηλωτές παραμένουν παρόντες. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργό ότι οι διαδηλωτές συνεργάζονται με τους τρομοκράτες, αυτό θα πρέπει να το εξηγήσουμε ότι δεν, μπορούμε να, δεν μπορεί να υποστηρίζει την Αραβική Άνοιξη, αλλά, δεν, αλλά να μην υποστηρίζει τη δημοκρατία και να μην την προστατεύει στην χώρα του. Χρειάζεται λοιπόν να εκφράσουμε και τη δικό μας αποτροπιασμό για το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης, τα κύρια μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία για τρεις μέρες δεν έκαναν καμία κάλυψη των γεγονότων. Τέλος όμως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας επιχειρηματολογία για να εμποδίσουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτήν την διαδικασία για να μπλοκάρουν τις προσδοκίες τη Τουρκία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο κύριος μαγνήτης για την Τουρκία η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι αυτοί που αγανακτούμε για αυτά που γίνονται στην Τουρκία αγανακτούμε γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η καλύτερη διαφύλαξη εναντίον τέτοιων αντιδημοκρατικών ενεργειών που είδαμε στην Τουρκία που πρέπει να πάψουν και μια για πάντα εκεί. Ο κύριος Νταφ, κύριε Πρόεδρε, με κάθε σεβασμό Απέναντι σε αυτά που είπε ο Τζαρ Πότμεν θα ήθελα να πω ότι η δήλωση της Άστον ήρθε αργά και δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και είναι εκτός περιεχομένου ουσιαστικά. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Τουρκία είναι μια δημοκρατική μορφή αφύπνισης Νομίζω ότι μπορούμε να τα συγκρίνουμε με αυτά που συνέβησαν στο Παρίσι το 1968. Δεν ήταν τα πάντα καλά τότε, δεν ήταν τα πάντα ειρηνικά και δεν ήταν τα πάντα δημοκρατικά. Αλλά όμως γνωρίζουμε ότι τελικά το 1968 άξιζε τον κόπο. Οι διαμαρτυρίες αυτές εκφράζουν λοιπόν μια μεγάλης διάρκειας δυσφορία και την ανικανότητα της πολιτικής ε, ηγεσίας της Τουρκίας να μπορέσει να αντικατοπτρήσει με σωστό τρόπο την τουρκική κοινωνία. Και υπάρχει και σύγκρουση ιδεολογιών από τη μία ο κεμαλισμός και από την άλλη το Ισλάμ. Κάτι το οποίο δεν βοηθά την δημιουργία μιας προοδευτικής φιλελεύθερης χώρας. Οι διαμαρτυρίες αυτές λοιπόν είναι ευρωπαϊκή θα έλεγα καταγωγής με την έννοια ότι είχαν συμβεί στην Ευρώπη πολλές φορές και θα πρέπει και η τουρκική κυβέρνηση να μάθει να σέβεται την έλλειψη κονφορμισμού και την έκφραση διαφωνίας. Νομίζω ότι μία από τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι να σταματήσει η προσπάθεια του Ερντογάν να γίνει υπερπρόεδρος στα πλαίσια ενός υπερπροεδρικού καθεστώτος. Thank you, President. Uh, let me start first. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τα βασικά συμπεράσματα για το τι συνέβη στην Τουρκία τις τελευταίες μέρες ένα δραματικά οικονομικό μπουμ, μια ανάπτυξη σε σχέση με τα προβλήματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπίεση της ελευθερίας έκφρασης οδηγεί σε εκρήξεις. Η ομάδα μου έχει επαναλάβει συχνά ότι η κυβέρνηση Ερντογάν συστηματικά δεν σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να σύλλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αν δεν υπάρξει πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχει ευρωπαϊκό μέλλον για την Τουρκία. Και δεν έχει μέλλον και σαν πρότυπη χώρα για την περιοχή, ένα ρόλο που θα ήθελε να έχει. Ο Ερντοάν με τη συμβολική που εκπροσωπεί και με τον ε, τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε την εξουσία πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, κατέστηλε βία τις διαδηλώσεις. Θα πρέπει με ταπεινοφροσύνη να δεχθεί να ζητήσει συγγνώμη. Για μας σοσιαλδημοκράτες το κίνημα ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και αυτή τη στιγμή ε, επεκτάθηκε σε όλη την Τουρκία και αυτό ήταν μια φόρμητη μορφή έκφρασης του τουρκικού πληθυσμού και δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόμμα που θα πρέπει να το διεκδικήσει. Πρέπει λοιπόν και εμείς εδώ να κατανοήσουμε το μήνυμα του τουρκικού λαού. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Λυπάμαι αλλά θα πρέπει και εγώ να, να συμφωνήσω με την ε, κυρία Ρόιτεν όπως επίσης και με τον κύριο Νταφ σχετικά με την καθυστερημένη αντίδραση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι είναι κάπως ενωρίς για να κριθεί οριστικά τι σημαίνει αυτή η διαμαρτυρία, η εξέγερση και η σύγκρουση. Όμως τα στοιχεία της, τα οποία προκύπτουν, μας δίνουν την ευκαιρία να τοποθετηθούμε. Και νομίζω ότι αυτό έκαναν και οι συνάδελφοι και κυρίως η εισηγήτρια. Ε, είναι ολοφάνερο ότι η Τουρκία ε, διανύει μια εποχή διεύρυνσης ε, των δυνατοτήτων της, ανάπτυξης όπως χαρακτηρίζεται από το διεθνές σύστημα, αλλά ταυτόχρονα μεγάλων δημογραφικών αλλαγών. Η Τουρκία έχει 15 εκατομμύρια φοιτητές, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή, στα πανεπιστήμια της και καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει. Αναδεικνύεται λοιπόν μια καινούρια μεσαία τάξη επιστημόνων οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καμία διάθεση επιστροφής σε, Ισλαμικού, σε Ισλαμικά δεδομένα αλλά υποθέτω ότι προφανώς δεν έχουν και καμία διάθεση να ζήσουν κάτω από όσα προσέφερε το κεμαλικό καθεστώς υπό την έννοια της αυταρχικής διακυβέρνησης. Ε, συμφωνώ και εγώ ότι είπα ότι εκπρόσωπος ε, καθυστέρησε να αντιδράσει. Ε, οφείλουμε να παρακολουθήσουμε στενά την υπόθεση αυτή διότι μπορεί να καταλήξει ε, σε πολύ μεγάλη σύγκρουση που δεν έχει σχέση βέβαια με την Αναβική Άνοιξη και ασφαλώς ένα μέρος αυτής της υπόθεσης οφείλεται στην τρέλα του μεγαλείου αν θέλετε κύριε Πρόεδρε στις ιδέες μεγαλείου που αναπτύχθηκαν διότι ο κύριος Ερντογάν και το κόμμα του έμεινε χωρίς αντίπαλο. Και βέβαια στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο κόμμα πολιτεύεται με τρόπο α, ιδιόρυθμο σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη προσεγγίζοντας σε προσωπικό επίπεδο τα άτομα, τις οικογένειες, δημιουργώντας συστήματα βοήθειας κτλ. τα οποία είναι ξένα προς την πολιτική πρακτική των δημοκρατικών χωρών. Ε, επομένως κύριε Πρόεδρε ε, ας είμαστε εν αναμονή αλλά σίγουρα αυτό είναι βέβαιο ε, κάτι δεν πάει καλά στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω και εγώ ότι δημοκρατία υπάρχει στα κράτη μόνον εφόσον υπάρχει απόλυτος σεβασμός της μειοψηφίας. Χωρίς απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος έκφρασης στη μειοψηφία δεν υπάρχει δημοκρατία. Χαίρομαι γιατί ακούω συνάδελφους ευρωβουλευτές οι οποίοι στο παρελθόν ε, μέρα νύχτα μας έλεγα για την Τουρκία που είναι το μοντέλο για τις δημοκρατίες της περιοχής πάρα πολύ γρήγορα είδαν την διαφαινόμενη αλλαγή και έστρεψαν την ανάλυση τους προς τη σωστή κατεύθυνση. Το τρίτο που έχω να πω είναι ότι η φράση της κυρίας Σόουμεν νομίζω ότι καθορίζει πλήρως την εικόνα της Τουρκίας. Έχει πει η κυρία Ομέν ότι η λέξη compromise δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της τουρκικής πολιτικής. Προχθές κύριε Πρόεδρε συμμετείχα σε διαδήλωση Τούρκων εδώ στις Βρυξέλλες για τα τεχτενόμενα στην Τουρκία. Μίλησα στους παρευρισκόμενους και τόλμησα να πω ως Κύπριος ότι παρότι μπορεί ό,τι πω να παρεξηγηθεί, εν τούτης του είπα δεν υπάρχει δημοκρατία στην Τουρκία αν στον αγώνα σας δεν ενταχθεί η υποχρέωση της Τουρκίας να αποσύρει τα στρατεύματά της από ξένα κράτη στα οποία υπάρχουν. Και χειροκροτήθηκα. Νομίζω ότι κάτι γεννιέται στην Τουρκία. Εμείς δεν κοιτάζουμε την Τουρκία από μια σκοπιά εχθρική καθόλου. Είμαστε υπέρ του τουρκικού λαού. Είμαστε αριστεροί προοδευτικοί άνθρωποι. Η έγνοια μας είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Και υποστηρίζομαι αυτή την έκρηξη ως μια νέα κατεύθυνση ε, των πολιτών της Τουρκίας. Νομίζω πως και αυτό που έχει πει ε, ο συνάδελφος ο κύριος Ταφ που έκανε σύγκριση με τον Μάη του 1968 ε, έχει εδώ ε, την θέση του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρος. Okay, well, thank you. Um, so, uh, Ευχαριστώ, λέει κύριος Στάνουκ. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόμα της ομάδας μου συμφωνώ με όλους αυτούς που λένε ότι δυστυχώς καθυστέρησε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να εκφράσει τις θέσεις της. Αυτοί που με ξέρετε δεν θα, δεν θα εντυπωσιαστούν όταν πω ότι πράγματι για πολλούς ε, λόγους υπήρξαν ε, αναδυόμενες εντάσεις δημογραφικές και άλλες στην Τουρκία τα τελευταία δέκα χρόνια. Αλλά η πλατεία Ταξίμ δεν είναι η πλατεία χρήματα και υπήρξε πράγματι υπερβολική βία που χρησιμοποιήθηκε από τις αστυνομικέ αρχές. Αν σκεφτούμε την, ιστορία της Τουρκίας τα προηγούμενα χρόνια, η αστυνομία πάντα είναι ιδιαίτερα επιθετική στην καταστολή των διαδηλώσεων και υπάρχουν βασικές ε, αντιπαραθέσεις σε σχέση με το μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει η Τουρκία στο μέλλον, αν θα πρέπει να είναι κοσμικό, θρησκευτικό, κεμαλιστικό, μετακεμαλιστικό και δεν πρέπει να μας εκπλήσει η συμπεριφορά του κυρίου Ερντογάν. Πριν από μερικά χρόνια ήθελε να ποινικοποιήσει την μοιχεία και τώρα το ε, αλκοόλ. Ενώ η χώρα, η χώρα του εισάγει σημαντικές ποσότητες ουίσκι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το επιτρέψει μόνο για ιατρικούς λόγους. Αλλά σίγουρα ο Ερντογάν είχε προτείνει το τουρκικό μοντέλο για την Αραβική Άνοιξη, για την Αίγυπτο κτλ. Τώρα θα πρέπει να καταλάβει τι θα πει να διαμαρτύρεται ο λαό όταν δεν είναι ικανοποιημένο με την ε, κυβέρνηση. Όταν λέει ότι όλοι αυτοί που πίνουν είναι αλκοολικοί, αυτό δεν έχει βοηθήσει την κατάσταση. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι θεωρεί ότι μόνος του πρέπει να αποφασίζει τα πάντα, ότι υπάρχει λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης, υπάρχει μια διαδικασία επικυριαρχίας του ΑΚΕΠΕ στην πολιτική και την οικονομία, αργά ή γρήγορα όλα αυτά θα οδηγούσαν σε διαμαρτυρίες. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι μαζί με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία φαίνεται ότι η Τουρκία ενισχύει και εξοπλίζει τους αλαφιστές στη Συρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ενισχυτικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και πρέπει να το καταδικάσουμε, να παρακολουθήσουμε τα θέματα πάρα πολύ προσεκτικά και να συνεχίσουμε να επικρίνουμε την τουρκική κυβέρνηση όταν δρά αντιδημοκρατικά και όλα αυτά θα πρέπει να φαίνονται και στην ετήσια έκθεση προόδου της Τουρκίας προς την κατεύθυνση της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Παρακαλώ να μην ξεπερνάτε το 1,5 λεπτό. Η κυρία Μουνής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε για το τουρκικό μοντέλο προκειμένου να εξαφθεί. εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα μάλλον ε, το μουσουλμανικό μοντέλο αρχίζει να εισάγει η Τουρκία και όχι το αντίθετο. Η κυρία Άστον Όντω, ίσω να άργησε, να καθυστέρησε, αλλά δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στην κυρία Άστον. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Εδώ και χρόνια έχουμε διαπραγματεύσει με την Τουρκία για τη διαδικασία ένταξη τη χώρα, η διεύρυνση τέλο πάντων τη Ένωση, με τα κεφάλαια 23 και 24 για τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν έχουν ανοίξει. Η Τουρκία είναι η χώρα όπου βρίσκονται περισσότεροι δημοσιογράφοι στη φυλακή από οπουδήποτε αλλού στην περιοχή και τις χώρες οι οποίες έχουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν δεν συγκρίνεται η Αραβική Άνοιξη με τόσα συμβαίνουν στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι δημοκρατία ενώ οι άλλες χώρες δεν ήτανε, ή επειδή στην Τουρκία υπάρχει οικονομική ανάπτυξη που δεν υπήρχε σε άλλες χώρες, αυτό που μπορούμε να συγκρίνουμε είναι την αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει και να αντιδράσει σε σχέση στα πλαίσια δηλαδή αυτής της διαπραγμάτευσης που κάνουμε και να επικεντρωθούμε στα κεφάλαια εκείνα που δημιουργούν πρόβλημα. Ο εξισλαμισμός είναι σοβαρό πρόβλημα. Όχι γιατί δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή βρετανικού ουίσκι στη χώρα, αλλά για άλλα προβλήματα πολύ πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα με την παραβίαση δικαιωμάτων γυναικών και άλλων μειονοτήτων. Ευχαριστώ. Ο... Σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλουμε να καταδικάσουμε καθαρά, χωρίς μισόλογα, την απαράδεκτη, βίαιη και προκλητική συμπεριφορά του Ερτογά και της κυβέρνησης του κατά του τουρκικού λαού, κατά της δημοκρατίας. Οφείλουμε να εκφράσουμε τη λύπη μας, την συμπάθεια και την αλληλεγγύη μας σε όλους εκείνους που έχασαν την ζωή τους, φυλακίστηκαν παράνομα, χτυπήθηκαν απάνθρωπα βία διαφωνώ και καταθέτω έντονα την απογοήτευσή μου, την διαμαρτυρία μου και την διαφωνία για τις μεθόδους που βία χρησιμοποιήθηκαν κατά πολιτών που είχαν κάθε δικαίωμα να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, την αντίθεσή τους για τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες. Η πλατεία Ταξίμ θύμισε τα πλατεία Ταχρή. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αποδεκτό, έστω ανεχτό από μια χώρα που θέλει να βρεθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια, να αντιμετωπίζει με νόμο το φιλί ως προσβολή της δημοσία εδούς. Πώς είναι δυνατόν με δρακόντιο νόμο να απαγορεύει το αλκοόλ. Πώς είναι δυνατόν να απαγορεύει στις αεροσυνοδούς των τουρκικών αερογραμμών να βάφουν τα χείλη και τα νύχια. Δεκάδες εκατοντάδες δημοσιογράφοι να φυλακίζονται. Να φημώνονται ουσιαστικά, να φημώνεται ουσιαστικά η ελευθερία του τύπου. Πώς είναι δυνατόν την ώρα των διαδηλώσεων σε περισσότερες από 67 πόλεις όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μεταφέρουν τη ροή της οφειλόμενης πληροφόρησης και το CNN Turk να προβάλλει σόου μαγειρική. Πώς είναι δυνατόν ο Σεβάν Νισανιάν Αρμένιος διανοούμενος να φυλακίζεται 13 μήνες επειδή άσκησε κριτική στον προφήτη Μουάμερ. Ο ίδιο το Σαΐν να φυλακίζεται σε 10 μήνες ο γνωστός μουσικός γιατί έκανε ένα αστείο Sir, σε ένα τμήμα, Κλείνω να πω ότι σήμερα πρέπει να καταδικάσουμε την απαράδεκτη κυβερνητική συμπεριφορά του Ερτογάν. Sorry, I did... Η κυρία Σάκη, ναι, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Θέλω να προσθέσω τη φωνή μου και σε αυτούς οι οποίοι είπαν ότι καθυστέρησε η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να αντιδράσει. Άκουσα τα σχόλια αυτά αν αποδειχθεί η, η ευθύνη της αστυνομίας τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει εμείς τώρα να καθυστερούμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Όλα αυτά είναι μια ευκαιρία να ξυπνήσει ο Ερντογάν και το ΑΚΕΠΕ και να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια στην αλαζονία της εξουσίας και την αυταρχικότητα. Η δημοκρατία δεν είναι μονάχα οι εκλογές και όποιος κερδίζει κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξυπνήσει, γιατί πολλές φορές νιώθω έλλειψη υποστήριξης όταν μιλάμε για την ανεξαρτησία των δικαστικών, το κράτος δικαίου, τις δίκαιες δίκης, τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ πιθανό ότι η πόλωση η οποία σοβεί στην τουρκική κοινωνία είχε πολλές φορές παραγνωριστεί γιατί θέλαμε να υπάρξει ένα μοντέλο οικονομικό και πολιτικό που θα ήταν φάρος σε μια δύσκολη περιοχή. Ο Επίτροπος κ. Φίλε πηγαίνει σε μια ήδη προβλεπόμενη συνδιάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη με οικοδεσπότη την τουρκική κυβέρνηση. Αλλά γιατί δεν, δεν ακύρωσε την παρουσία του και δεν πήγε να, έχει, να ζητήσει από την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τη βία της αστυνομίας και να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα και να περάσει απλώς λεκτικές ε, διατυπώσεις και να εστιάσει στην κοινωνία των πολιτών και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στο διαδίκτυο και στον έντυπο ε, Γιατί λοιπόν δεν σταματάμε τις εξαγωγές ε, δακρυγόνων στην Τουρκία αν καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές. Δεν περίμενα αυτή τη στιγμή για να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει την προσχώρηση της Τουρκίας. Πρέπει να σκεφτούμε και πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε σε διάλογο με την Τουρκία για να γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή όλων των πολιτών στην Τουρκία. Και εδώ το ΕΛΚ μπορεί να κάνει κάτι, γιατί το ΑΚΕΠ είναι παρατηρητής στην Ένωση των Χριστιανοδημοκρατών. Εντάξει. Πρέπει να κάνει κάτι το ΕΛΚ για όλα αυτά. Κυρία Θεοχάρους. Ακούσαμε σήμερα δύο ψυχαναλυτικέ ερμηνείε τη κατάσταση στην Τουρκία, μια από την κυρία Γιαννάκου που είναι ψυχίατρο, μια από τον κύριο Τάνοκ που είναι ψυχίατρο, αλλά ακούσαμε και μια από την Κομισιόν, η οποία μέσα από μια βελούδινη προσέγγιση προσπάθησε να μα πείσει ότι η εξέγερση του λαού τη Τουρκία δεν έχει καμιά σχέση με την εξέγερση σε ολόκληρο τον κόσμο σε άλλου μουσουλμανικού λαού. Εκείνο που έχει πετύχει η Κομισιόν είναι να μα πείσει ότι εκείνο που μετράει είναι ο όγκο των συναλλαγών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία είναι η στρατηγική της θέση και όχι οι αρχές και οι αξίες και η δημοκρατία για την οποία κόπτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πολλοί δεν βλέπουν εκείνο που βλέπει όλος ο κόσμος, δηλαδή την ε, κρυφή, την προσωπική ατζέντα του Ερτογάν να οδηγήσει τη χώρα να διολυστήσει προς τον Ισλαμισμό. Ανεγείρονται παντού τζαμιά, μιναρέδες, Ισλαμικά σχολεία. Δυστυχώς αυτό έχει συμβεί και στην κατεχόμενη πατρίδα μου. Δυστυχώς εκεί βιάζεται το γαλήνιο τοπίο της κατεχόμενης Κύπρου με όλα αυτά που κάνουν. ιστορίες με το αλκοόλ, με τον οικογενειακό προγραμματισμό, πόσα παιδιά θα κάνει ο καθένας, η καταστολή του ίντερνετ, τα Ισλαμικά σχολεία όπως έχω πει, όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία ξεφεύγει από τον δρόμο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Παράλληλα, είναι και ο ηγεμονικός ρόλος τον οποίο επιδιώκει να παίξει ο Ερτογάν και η Τουρκία σαν μοντέλο για τους υπόλοιπους α, αραβικούς Ισλαμικούς λαούς και νομίζω, τελειώνω Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, ε, ε, ελάχιστες φορές μου δίνετε το χρόνο, Όποιο θέλει, όποιος θέλει να βοηθήσει την Τουρκία. Ε, ο Κύριος Κουμουτσάκος αν δεν έχουμε πειθαρχία, τότε δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, δεν θα μπορέσουμε όλοι να λάβουμε. Είμαι εδώ από τις 9 η ώρα, λέει η κυρία Θεοχάρη, για να λάβω το λόγο. 1,5 λεπτό για όλους. Έχουμε τέσσερις ομιλητέ. Και έχουμε μετά την ακρόαση του πρεσβευτή που περιμένει. Παρακαλώ. Κύριος Κουμουτσάκος. But it's also sorry when I would like to say, talk to your colleagues who have not και μιλήστε στους συναδέλφους που δεν έχουν περιοριστεί στο 1,5 λεπτό, αν έχετε διαμαρτυρίες. Χρειάζεται πάντα να υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ μας. Πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες για να έχουν όλοι τον χρόνο να μιλήσουν. Κύριο Κουμουτσάκος. Τα δραματικά και δυστυχώς αιματηρά γεγονότα στην Τουρκία έχουν εμφανείς αφορμές. Όμως οι ρίζες και οι πραγματικές αιτίες τους είναι βαθιές και σοβαρές. Η αναστάτωση στην οποία βρίσκεται η τουρκική κοινωνία και η Τουρκία σήμερα δεν είναι παροδικό φαινόμενο. Φοβάμαι ότι είναι σταθερό χαρακτηριστικό που θα επανέρχεται όσο η αναζήτηση σαφούς εθνικής ταυτότητας και εθνικού προσανατολισμού αυτής της χώρας συνεχίζεται. Όσο η σκληρή διελκυστίνδα μεταξύ κοσμικής, λαϊκής και θρησκευτικής Τουρκίας, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, δεν έχει σταματήσει. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η ευρωπαϊκή προοπτική τη Τουρκία δεν έχει κρυθεί. Όχι γιατί η Ευρώπη δεν έχει τηρήσει τι υποσχέσει τη, όπω συνηθίζουν να λένε και να ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι του τουρκικού κράτου, αλλά για... γιατί η Τουρκία, όπω φάνηκε αυτέ τι μέρε, δεν μπορεί να αποφασίσει ακόμα, εάν θέλει και μπορεί, να ακολουθήσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τον ευρωπαϊκό δρόμο και τι υποχρεώσει που αυτό ο δρόμο συνεπάγεται και πρωτίστως όσον αφορά τη θεμελιώδη αρχή του σεβασμού των ανθρωπίνων και ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, το σεβασμό και την υποχρέωση δημοκρατικής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει Κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ζήτησα το λόγο κυρίως ε, να καταγγείλω την απαράδεκτη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα γεγονότα στην Τουρκία. Είναι απαράδεκτο αυτό που ακούσαμε και τώρα. Ακούστηκε από τον εκπρόσωπο της ε, κυρίας Άστον ότι θα τα καταδικάσει η Ένωση εάν αποδεχτούν οι κατηγορίες. Μα τα δαμε όλοι μας. Τι άλλο να περιμένει ας πούμε. Και για μας υπάρχει η εξήγηση γιατί υπάρχει αυτή η θέση και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια πλευρά να, να χειροκροτεί την Τουρκία για το ρόλο της στη Συρία δεν μπορεί να χειροκροτεί για το ότι φιλοξενεί δεν ξέρω πόσε συναντήσει των αντικαθιστοτικών στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μπορεί να τη χειροκροτεί για το ότι έχει εγκαταστήσει του Patriot και από την άλλη μεριά να, να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Είναι ε, απαράδεκτη αυτή η στάση. Ακούστηκαν διάφορε αναλύσει. Αυτό που δεν υπόθηκε από κανέναν είναι το γεγονό ότι αυτή η εξέγερση αντικατοπτρίζει και μια άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Τούρκοι εργαζόμενοι. Με πολύ χαμηλού μισθού, με μια παράδεκτη κατάσταση όσον αφορά τι εργασιακέ σχέσει, με φτώχεια, ανεργία και περιθωριοποίηση. Και το γεγονό ότι τα, και τα συνδικάτα, αυτά τα ελεγχόμενα συνδικάτα μπαίνουν στον αγώνα, δείχνει ακριβώ την, την έκταση που έχει αυτή η, κατάσταση. Και εμεί είμαστε πλήρω αλληλέγγυοι με τον αγώνα των Τούρκων εργαζομένων, αλληλέγγυοι με τον αγώνα του Κομμουνιστικού κόμματο Τουρκία, το οποίο θρυνεί θύματα συλλήψεις και καταστροφές και πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας δεν θα σταματήσει γιατί πλέον οι εργαζόμενοι ξέρουν ποιο είναι το δίκαιό τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα τρία πιο ανησυχητικά πράγματα είναι η ανταπόκριση της αστυνομίας, η αποτυχία της τηλεόρασης να καλύψει τις ταραχές και η καταδίκη από τον Πρωθυπουργό αυτών που χρησιμοποιούν τα, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Δεν αμφισβητείται εδώ η νομιμότητα του κράτους, αλλά εκφράζεται μία δυσφορία μία δυσφορία ανάμεσα και σε αυτούς που ψήφισαν το ΑΚΠ γιατί θεωρούν ότι το ΑΚΠ περιφρονεί την κοινή γνώμη παρότι υποτίθεται το κόμμα αυτό οδηγεί την Τουρκία στην πρόοδο, αλλά το κόμμα αυτό είναι ένας συνασπισμός τελικά διαφορετικών δυνάμεων και βλέπουμε ότι ίσως να σπάσει ανάμεσα σε ένα κομμάτι προοδευτικό φιλελεύθερο και ένα κομμάτι συντηρητικό ισλαμικό. Αν κάτι τέτοιο γίνει δεν θα είναι καλό για την Τουρκία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που δεν άκουσα εγώ είναι ένα ισχυρό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρόκειται βέβαια για το τι χρώμα θα είναι το κραγιόν, αλλά πρόκειται για τις βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες που εδώ, εδώ και χρόνια ε, καταδικάζουμε την έλλειψή τους. Είναι το θέμα της συμπεριφοράς της αστυνομίας. Είναι η έλλειψη ελευθερίας του τύπου. Το σημαντικό εδώ, αν θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα, είναι να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα με την Τουρκία, όσο γίνεται πιο γρήγορα όπως το έχουμε πει συχνά. Και να φροντίσουμε να είναι σαφές για την Τουρκία το τι συμβαίνει και τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει βελτίωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι... Σας ευχαριστώ Πρόεδρε θα θέλαμε να πούμε το εξή. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν την προσέγγιση με την Ευρώπη και αυτών που είναι συντηρητικοί και οι οποίοι είναι η κύρια πηγή στήριξη στο καθεστώς του κυρίου Ερντογάν. Αυτό είναι ένα τμήμα της κοινωνίας. που είχαν διεκδικήσει και στο παρελθόν την εξουσία στην Τουρκία. Δεν πρέπει λοιπόν να διακόψουμε τους δεσμούς που έχουμε με την Τουρκία. Αντίθετα, στο φως των νέων εξελίξεων στην Τουρκία, νομίζω ότι μπορεί να προκύψει μια νέα σύνθεση, μια νέα μορφή συμβιβασμού και υπάρχει και η ευκαιρία να επιληθεί το κουρδικό στην Τουρκία σήμερα. Αυτό είναι ένα μια ένδειξη ότι υπάρχει θέληση για διάλογο. Πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24 με την Τουρκία, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στην Τουρκία, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και αυτό θα ήθελα να ζητήσω από του συναδέλφου να ανοίξουμε αυτά τα κεφάλαια. Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πέρα από την απάντηση, το αν έγινε γρήγορα ή αργά από πλευράς της κυρίας Άστον, πρέπει να αντιληφθούμε το εύρος των ε, γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σήμερα στην Τουρκία. Το θέμα της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας του τύπου. Τίποτα δεν θα ήταν πιο σοβαρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα συμφέροντά της από μια αποσταθεροποίηση της Τουρκίας έτσι όπως τη βλέπουμε και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι μια υπεύθυνη απάντηση με συνέπεια απέναντι στις αρχές και τις αξίες μας. Μια σταθμισμένη απάντηση, μια απάντηση που να μην είναι δυσανάλογη και που να μην ευνοεί αστάθεια, όπως είπαμε πριν, για να μην οδηγηθούμε εκεί όπου έχουμε οδηγηθεί και σε άλλες χώρες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Συνοχή με τις αξίες και τις αρχές μας, και να έχουμε μια σε βάθος συζήτηση για το τι συμβαίνει στον αραβικό κόσμο, ο εξισλαμισμός δηλαδή των κοινωνιών και κατά πόσο τηρούν ή όχι ανθρώπινα δικαιώματα οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. οι Κομισιόν θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ενημερώσω για το ότι ο Επίτροπος Φίλε στην Κωνσταντινούπολη δεν θα συναντηθεί μόνο με τον Πρωθυπουργό Ερτογκάν και τον Υπουργό Βάκης, αλλά και με την πλατφόρμα του Ταξίμ και με ε, την κοινωνία των πολιτών. Ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι οι αρχές έχει υποστηρίξει μέχρι τώρα και με τον ίδιο τρόπο θα τις υποστηρίξει και αυτή τη φορά στην Τουρκία. Hello. They do not understand. So, thank you very much for this. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συζήτηση αυτή. Ήταν μια έντονη και σημαντική συζήτηση και θέλω να περάσω τώρα στο επόμενο σημείο και κλεισμένων των θυρών γιατί χάσαμε πολύ χρόνο. Not lost. We used the time for other purposes. Χρησιμοποίησαμε το χρόνο για άλλους στόχους πρέπει να κάνουμε γρήγορα και γιατί έχουμε δύο ακόμα σημεία να διεκπαιρεώσουμε.